προς μια ε, θετική ψήφο αυτή την πρόταση αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, έχει κλείσει η συζήτηση στο θέμα αυτό. Αύριο ψηφοφορία στις 11.30. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο. Πρόταση ψηφίσματος, τεχνικές απαιτήσεις και διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά τις πτυτικές λειτουργίες. Εκ μέρου τη Επιτροπή Μεταφόρων και Τουρισμού θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Μπράιαν Σίμψον να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Ως πρόεδρος της Επιτροπής έπρεπε εγώ να υποβάλω επίσημα το ψήφισμα που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού και που απορρίπτει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το χρόνο πληρώμα πτήσεων και υπηρεσίας. Οι προσωπικές μου απόψεις διαφέρουν λίγο από εκείνες που υιοθέτησε τότε η Επιτροπή, αλλά παρόλα αυτά σας υπο, υποέβαλα ε, και τυπικά αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Επίτροπος Καλάς. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η πρόταση της Επιτροπής για τους περιορισμούς, τους χρόνους πτήσης δεν είναι μια τυπική νομοθετική πρόταση, είναι κανονισμός ασφαλείας. Εγκρίθηκε από την Αρμόδια Ρυθμιστική Επιτροπή των Κρατών Μελών στις 12 Ιουλίου του 2013 με συντριπτική πλειοψηφία. Ο Ευρωπαϊκή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας ε, κλήθη να εκπονήσει κανόνες ασφαλείας για την αεροπορία. Προσωπικά πιστεύω ότι τα, οι λεπτομέρειες του κανονισμού ασφαλεία δεν θα πρέπει να τίθενται σε πολιτική συζήτηση. Θα πρέπει να υπάρχουν οι εντεταλμένοι, εξουσιοδοτημένοι ειδικοί που θα τα συζητήσουν αυτά. Όταν διαπραγματευόμεθα με τους ε, τέρους μας στο εξωτερικό και είχαμε πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα με χώρες ε, στην Ανατολή και τον Νότο, ε, Οι εταίροι μας με τους οποίους διαπραγματευόμαστε λένε ότι οι πολιτικές παρεμβάσεις πρέπει να αποκλείονται. Για να διευκολύνουμε την επικοδομητική λήψη αποφάσεων θα ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις για τον κανονισμό αυτό. Πρώτον, εις ό,τι αφορά το σημείο 5 στις πρώτες της Κομισιόν τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόσουν και να επιβάλλουν στις αεροπορικές εταιρείες διατάξεις πιο προστατευτικές από αυτές που προβλέπει ο κανονισμός ε, με την πρόθεση ότι το αίτημα του κράτους μέλους έχει ε, τύχει της σωστής επεξεργασίας και καλύπτονται ή ξεπερνώνται τα πρότυπα ασφαλείας. Δεύτερον, οι ενωσιακοί κανόνες για το stand-by ε, έχουν διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο το, ώστε να μην είναι κανείς περισσότερο ε, σε υπηρεσία ε, από 18 ώρες. Επίσης θα πρέπει οι διατάξεις ασφαλείας να είναι διατυπωμένες έτσι ούτως ώστε κανείς να μην είναι σε υπηρεσία μετά από 18 ώρες. Εις ό,τι αφορά τις νυχτερινές πτήσεις, η Κομισιόν θα ζητήσει από την ΕΑΣΑ, την Υπηρεσία Ασφαλείας, να συμπεριλάβει ε, στις προδιαγραφές πιστοποίηση ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα εφαρμόζουν ε, ε, σχέδια διαχείρισης της κόπωσης όταν υπερβαίνει η διάρκεια τη πτήσης τις 10 ώρες τη νύχτα. Επίση, οι εμπλεκόμενοι, συμπεριλαμβανομένοι των εκπροσώπων των πληρωμάτων, θα παραμένουν και θα εξακολουθούν να συμμετέχουν ε, σε όλες ε, τις εξελίξεις αυτού του θέματος, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει ή όχι την προτινόμενη νομοθεσία και να διατηρήσει για αρκετά χρόνια ακόμα τους εθνικούς κανόνες. Ο χρόνος πτήσης δεν είναι μη ρυθμισμένο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σεβαστεί την όποια απόφασή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω τώρα τον κύριο Κρός να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, δύο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω συγκεκριμένα εκείνους που ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα που από τεχνικής πλευράς δεν είναι καθόλου απλό όσους συνέβαλαν να, ώστε να έχουμε σωστή πληροφόρηση εδώ στο Κοινοβούλιο, ούτως ώστε να μπορούμε να στηρίξουμε ένα σωστό νομοθέτημα. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Σάιντλ Κατραβή, ο οποίο προσπάθησε να διευκρινίσει τα σκοτεινά σημεία μέχρι τελευταία στιγμής, ε, ούτω ώστε να απαντηθούν οι ερωτήσεις από όλε τις πολιτικές ομάδες. Και η τοποθέτηση του Επιτρόπου το έδειξε αυτό. Ω ε, ΕΛΚ ε, δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια και Κανέναν δεν αφήνουμε να μας επικρίνει ότι είμαστε το μακρύ χέρι της βιομηχανίας ή το μακρύ χέρι άλλων λομπιστών. Εμείς θέλουμε ασφάλεια για το προσωπικό και τους επιβάτες. Και όλα τα άλλα είναι λάθος και βεβαίως ε, μπορεί να αντιβαίνουν σε όλες μας τις πρωτοβουλίες. Η πρόταση της Κομισιόν μετά τις έρευνες που κάναμε και εμείς ε, αποτελεί οπωσδήποτε μία πρόοδο σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Ίσως δεν έχουν επιτευχθεί όλα όσα κάποιοι ανέμεναν, αλλά σίγουρα αποτελεί πρόοδο δεν νομίζω ότι είναι σωστό να πούμε ότι αποτελεί οπισθοδρόμηση. Αυτό είναι το σημαντικότερο επιχείρημα για να στηρίξουμε τη θέση της Κομισιόν. Οι διευκρινήσεις του Επιτρόπου απόψε σημαίνουν, κατά τη γνώμη μας επίσης, ότι αυτό που ρυθμίζεται με αυστηρότερο τρόπο στα κράτη-μέλη δεν αναιρείται και αυτό είναι πολύ σημαντικό και ε, ιδιαίτερα ε, τέτοια μέτρα ε, θα πρέπει να ρυθμίζονται διαδικαστικά με τους εμπλεκομένους. Οπότε και το τέταρτο σημείο είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζω ότι αντίστοιχα και στο μέλλον θα κάνουμε εδώ έναν αντικειμενικό διάλογο και όχι έναν διάλογο που διαστρεβλώνει την πραγματικότητα όπως έχει συμβεί πρόσφατα αρκετές φορές. Ευχαριστώ. Κύριος τρία λεπτά. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Ε, θα ήθελα να πω ότι γνωρίζω την πολυπλοκότητα του θέματος αυτού και τις δυσκολίες που ενέχονται όμως αν δούμε τα γεγονότα πρέπει να τα αξιολογήσουμε και να καταλήξουμε σε συμπέρασμα και θέλω να πω εδώ από την αρχή κάτι για τη διαδικασία υπήρξε μεγάλη κριτική σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε όμως είναι το αποτέλεσμα των κανονισμών που ενέκρινε αυτό το κοινοβούλιο. Πριν κάποιο χρονικό διάστημα είχαμε πει τότε ότι αυτά τα τεχνικά ζητήματα πρέπει να φεθούν στους εμπειρογνώμονες ότι για τρία χρόνια ε, εργαστήκαμε στο αυτό και τους τελευταίους εξή μήνες εργάστηκε σε αυτό το θέμα η Κομισιόν ε, και διαβουλεύτηκε και με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατόπιν ελήφθη μια απόφαση. Αυτή εγκρίθηκε από τους εμπειρογρόπονες των κρατών μελών και τώρα έχουμε αυτό το φάκελο και μπορούμε είτε να διταχθούμε είτε όχι. Αυτή είναι δική μας επιλογή. Τις τελευταίες εβδομάδες Ακούσαμε πάρα πολλά σχετικά με το φάκελο αυτό και ασκήθηκε κριτική. Εγώ είμαι σύμφωνος με κάποιες από τις κριτικές που έγιναν, όμως σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και το είπε και ο κύριος Σίμψον ότι αν κάνουμε αντικειμενικά τη σύγκριση μεταξύ αυτού που έχουμε τώρα επιτάπητος αφενός και αφετέρου ποιοι είναι σε σχέση με το ποιοι είναι οι διεθνείς κανόνες ασφαλείας, τότε στο 95% των περιπτώσεων καταλήγουμε με μια καλύτερη κατάσταση ή με μια κατάσταση ταυτόσιμη με τη σημερινή. δεν ε, θα πρέπει να συγκρίνουμε με το τι ισχύει στη θεωρία, αλλά το τι γίνεται στην πράξη σήμερα στα κρατη Εδώ Μιλάμε για συλλογικές συμβάσεις ε, και για μια σειρά άλλων πραγμάτων και δεν μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο καθεστώς ε, και είναι καλό που ακούσαμε τον Επίτροπο να επαναλαμβάνει απόψε ότι τα εφιστάμενα καθεστώτα είναι βασισμένα σε εργατική νομοθεσία και σε νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση και τελικά θα έχουμε περισσότερη ασφάλεια. Η ρήτρα της ε, μήνα είναι ένα σημαντικό θέμα και οι 18 ώρες, ο περιορισμός των 18 ώρων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά αποτελούν μια καλή βάση και μπορούμε να βασιστούμε στα επόμενα έτη για να οικοδομήσουμε κάτι καλύτερο και με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η δική μου συμβουλή λοιπόν είναι να μην ε, απορρίψουμε την πρόταση απόρριψης ε, και να υποστηρίξουμε την πρόταση της Κομισιόν ε, λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινήσεις που δόθηκαν. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε Καλάς για τις επεξηγήσεις σας. Δεν αντιμετώπισα ε, με ευκολία το θέμα. Ε, είχα τις επιφυλάξεις μου αν είναι σωστή η θέση αυτή ε, ή η θέση μας του 2008 για τη σύσταση ειδική επιτροπής και ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλισης Αεροπορίας. Είχαμε πολλές συζητήσεις, είχαμε την ακρόαση στην Επιτροπή Μεταφορών, μίλησα και με πολλούς πιλότους, ε, με πιλότους με το συνδικάτο τους. Και τέλος κατέληξα μετά από όλα αυτά ότι η πρόταση αυτή είναι συμβιβαστική λύση καλή και θα μπορούσε να υποστηριχθεί. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερη. Αναφέρομαι ε, ειδικά ε, στα θέματα που συζητήσαμε και στο hearing στην ακρόαση ότι δεν μπορεί να ξεπερνάει η νυχτερινή διάρκεια της πτήσης στις 10 ώρες. Στις ΕΠΑ είναι 9 ώρες. Ε, εδώ έχουμε 11 αντί για 11 και 45 που ήταν πριν. Είναι παραπάνω από τις 9 και παραπάνω από τις 10 ώρες. Αν συγκρίνουμε με τις ΕΠΑ έχουν πολύ πιο σύντομες, σύντομους χρόνους ανάπαυσης ε, μετά από διπυρωτικές πτήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι καλύτερα είναι να διατηρήσουμε τις 11 ώρες και να έχουμε μεγαλύτερο χρόνο ανάπαυσης μετά το χρονικό διάστημα της πτήσης. Πιστεύω ότι η πρόταση αυτή από πολλές απόψεις συνιστά σαφή βελτίωση σε σχέση με την τωρινή κατάσταση ε, που επικρατεί σε πολλά κράτη-μέλη και αυτό που είχαμε μέχρι τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και περί αυτού πρόκειται σε τελευταία ανάλυση. Ε, αναφέρθηκε επίση ότι αν ένα κράτο μέλο θέλει να τα κάνει ακόμα καλύτερα, να δημιουργήσει ακόμα καλύτερε συνθήκε ή και μία αεροπορική εταιρεία να το κάνει, δεν απαγορεύεται, αντίθετα επιτρέπεται. Το σημαντικό είναι ότι έγιναν μεγάλες πρόοδοι με την συμβιβαστική αυτή πρόταση. Στην αρχή δεν είχαν συμφωνήσει, δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδεις και οι αεροπορικές εταιρείες. Τώρα επίστησαν και ε, έχουμε βρει μια συμβαστική λύση για τις ε, προϋποθέσεις ασφαλείας. Τρία κράτη-μέλη ε, τώρα έχουν καλύτερα δεδομένα από τα δικά μας, αυτά που υπάρχουν στην πρόταση δηλαδή. Γι' αυτό η γνώμη μου είναι να απορριφθεί το ψήφισμα αύριο και να υποστηριχθεί η πρόταση κυρίως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν υποστηριχθεί το ψήφισμα αύριο, τότε θα έχει γίνει όλη η δουλειά επιματέω και σίγουρα το τελικό αποτέλεσμα θα είναι χειρότερο από αυτό που προβλέπει η πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και για δυόμιση λεπτά τώρα ο κύριος Κράμερ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το 2009 στο Μπάφαλο ε, υπήρξε μια τρομερή, ε, ε, ένα τρομερό αεροπορικό ατύχημα που κόστισε τη ζωή σε 50 ανθρώπους και οι δύο πιλότοι είχαν αποκοιμηθεί. Ε, στο μαύρο κουτί φαινόταν ότι κοιμόντουσαν και από τότε είχαν πει στη ΣΥΠΑ ότι 9 ώρες νυχτερινή πτήση και 16 συνολικά. Απέχουμε πολύ. Κάθε τρίτος πιλότος έχει ομολογήσει ότι τον έχει πάρει ο ύπνος και κάθε δεύτερος είπε ότι και ο ε, δεύτερος πιλότος αποκοιμήθηκε. Ε, δύο στη Βρετανία αποδεδειγμένα αποκοιμήθηκαν, αλλά ευτυχώς δεν συνέβη τίποτε. Και τώρα το... Η τωρινή πρόταση στηρίζεται στον κανονισμό 216 του 2008 που ε, ε, πρόβλεπε να ε, αποφασιστούν συγκεκριμένες χρονικές διάρκειες πτήσης. Δέκα επιστήμονες εξουσιοδοτημένη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας και τέσσερις άλλες μελέτες μιλάνε για δεκάωρο μάξιμουμ αλλιώς ε, διακυβεύεται η ασφάλεια. Αυτό πρέπει να είναι η κατευθυντήρια γραμμή. Γιατί μιλάτε για 11 ώρες, διότι από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική, τις ανατολικές ακτές χρειάζονται 11 ώρες και θα πρέπει να έρθει κι άλλος πιλότος εάν μειωθεί το όριο αυτό. Αυτό σημαίνει ε, ε, αύξηση 1,5 ευρώ ανά εισιτήριο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα υπάρχει άνθρωπος που θα πει δεν πληρώνω 1,5 ευρώ παραπάνω αλλά επί 11 ώρες θα τρέμω, μπας και αποκοιμηθεί κανένας πιλότος. Η ασφάλεια για τους ε, επιβάτες πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Τρία χρόνια δεν κινήθηκε τίποτα και λίγο πριν από τη συζήτηση έρχεστε εδώ με τρίμπλες για να διασφαλίσετε την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου που φοβάστε ότι δεν θα την έχετε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Τι ε, ε, θα γίνει αν ε, το ατύχημα του Μπάφαλο γίνει και στην Ευρώπη. οι, τουλάχιστον οι Αμερικανοί άλλαξαν τις διατάξεις. Αν γίνει ένα τέτοιο ατύχημα, εσείς θα είστε υπεύθυνος που δεν δεχτήκατε τις 10 ώρες Υπεύθυνοι θα είναι και εκείνοι οι συνάδελφοι αύριο που θα ψηφίσουν κατά του δικού μας του ψηφίσματος και υπέρ της δικής σας της πρότασης. Γι' αυτό σας παρακαλώ να ψηφίσετε υπέρ του δικού μας ψηφίσματος, ούτως ώστε να έχουμε ασφάλεια για τα πληρώματα και τους επιβάτες. Ευχαριστώ. Κύριε Κράμερ, θα δεχτείτε μια μπλε κάρτα από την κυρία Μάισνερ. Κυρία Μάισνερ. Αγαπητέ κύριε Κράμερ, Βεβαίω η ασφάλεια στις μεταφορές μας απασχολεί όλους, ιδιαίτερα ε, μας απασχολεί η ασφάλεια σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Όμως ε, η ασφάλεια ε, στους ε, ουρανούς δεν πιστεύετε ότι είναι υψηλή στην Ευρώπη. Αν ήταν τα πράγματα όπως τα παρουσιάσατε και έπαιρναν οι, πιλότοι, πολλοί πιλότοι τον υπνάκο τους, τότε τα ατυχήματα θα ήταν πολύ περισσότερα. Ε, μπορούν επίσης να πούν ότι, ε, να πει ένας πιλότος ότι δεν ε, μπορεί να αναλάβει την πτήση. Ναι, αλλά φοβάται ότι θα του καταγγείλουν τη σύμβασή του. Το ψήφισμα αντιμετωπίζει πολύ καλύτερα όλα αυτά. Οι προδιαγραφές πιστοποίησης είναι ένα άλλο θέμα επίσης. Δεν τις έχουμε δει, αλλά τις ψηφίζουμε και προβλέπουν 3,5 ώρες παραπάνω από αυτές που συζητούμε. Δεν είμαστε ενημερωμένοι. Ψηφίζομαι για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Επίσης θέλουμε νομοθετικό έργο για ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν μπορεί δηλαδή, γι' αυτό, αυτό είναι το δικό σας έργο κυρία Κάλασε. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις επιταγές και τις προτροπές της επιστήμης 10 ώρες. Ε, ε, Η κυρία Φώστερ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και Ενταμέλη. Εκ μέρου τη ομάδα μου είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη που βλέπω αυτό το ψήφισμα ενώπιον τη Ολομέλεια και ακόμη πιο απογοητευμένη από ένα ε, μεγάλο βαθμό παραπληροφόρηση γύρω από το θέμα αυτό. Έχω όλε τι πληροφορίε, κύριε Κράμερ, αν χρειάζεστε περισσότερες. Ε, δούλεψα ε, ως πλήρωμα τα πρώτα 25 χρόνια πρωτού γίνω ευρωβουλευτή και ασχολήθηκα με του περιορισμού χρόνου πτήσεως και πολλέ άλλε εργασιακέ συμφωνίε ω ε, διαπραγματεύτρια συνδικαλιστική. Η πραγματογνωμοσύνη μου σε αυτό τον τομέα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Σα ε, βεβαιώ ότι είμαι η τελευταία που θα λάβω ε, ελαφρά την καρδιά τα θέματα ασφάλεια, διότι ήμουν υπεύθυνη για την υποχρεωτική αναφορά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά άλλα θέματα. Για τέσσερα χρόνια περίπου τα συνδικάτα του κλάδου ε, και άλλοι εμπειρογνώμονες συμμετείχαν σε αυτές τις συζητήσεις μετά από εκτεταμένες έρευνες μαζί με τα τελευταία επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία που υπάρχουν οποιοδήποτε περιορισμοί και κανόνες χρόνου πτήσης θα πρέπει να θεωρηθούν ως ένα πλήρες πακέτο και όχι ως μια σειρά από μεμονωμένες απαιτήσει. Αυτό το πακέτο μέτρων περιέχει ε, ορισμένες διατάξεις που θα πρέπει να αφορούν βελτιώσεις ασφάλειας στον κανονισμό γενικά. Αυτές οι αλλαγές γενικά εφαρμόζουν πιο αυστηρούς κανόνες από αυτούς που υπάρχουν στις περισσότερες χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Για να είμαστε σαφείς, αυτός ο κανονισμός δεν έχει εντολή να επηρεάσει ε, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Είναι ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο έχει την ασφάλεια στο επίκεντρο. Οι πιο αποτελεσματικοί κανόνε θα εφαρμόζονται πάντοτε, διασφαλίζοντας ότι ε, ε, διασφαλίζοντας πάντα τα ύψιστα επίπεδα ασφάλεια. Εν κατακλείδη, η αρχή πολιτικής αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου και, όλων, και όλες οι αρχές των άλλων κρατών και οι κυβερνήσει των κρατών μελών υποστηρίζουν αυτή την αναθεώρηση και ελπίζω ότι θα απορρίψουμε αυτό το ψήφισμα. Ωστόσο, ε, θα εισηγόμουν ότι τα κόμματα ε, να αναφερθούν πίσω στην ε, Επιτροπή Μεταφορών ένα χρόνο μετά από την εισαγωγή των κανονισμών. Κύριε Πρόεδρε, προέρχομαι από ένα έθνο νησί που στηρίζεται σε έναν ασφαλή τομέα μεταφορών, ιδιαίτερα τον τομέα των αερομεταφορών, για τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών. Και θα θέλω να διασφαλίσω ότι όλοι οι επιβάτες μπορούν να ε, χρησιμοποιούν τις αερομεταφορές ε, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας και επιβάλλονται με αποτελεσματικότητα. Και γι' αυτό η ομάδα μου θα υποστηρίξει τον κανονισμό όπως εφαρμόζεται. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Αμπίλση. Για λεπτά. Ευχαριστώ. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τις, τους χρόνους πτήσης ε, πραγματικά είναι τελείως ανεύθυνες και υπονομεύουν την ε, ανθρώπινη ζωή. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή πότε θα γίνει ατύχημα επειδή έχουν υπερκόπωση οι πιλότοι. τώρα ε, ήδη ε, πολλές ε, ανομαλίες οφείλονται στην υπερκόπωση ή την κόπωση των πιλότων. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι κατά μέγιστο για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να υπερβαίνονται οι 10 ώρες. Τώρα εργάζονται πολύ περισσότερο. Μπορεί να είναι ένας πιλότος ξύπνιος 22 ώρες. Ο κουρασμένος πιλότος ε, δεν μπορεί να αντιδράσει σωστά. Η ασφάλεια των ε, επιβατών θα πρέπει να ε, είναι πάνω από τα κέρδη των αεροπορικών εταιριών. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Θα πρέπει να κάνουν οικονομίες για να αυξάνουν τα κέρδη τους. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν λαμβάνουν υπόψη ε, τέσσερις μεγάλες μελέτες ανεξάρτητων ειδικών. Η, η Κομισιόν επίσης ε, ανέβαλε τα μέτρα, ε, ορισμένα μέτρα ασφαλείας ε, για να αποφύγει το... και ε, ε, προχώρησε σε διαδικασίες εντοτικού δικαίου για να, μην... για να αποφύγει την παρέμβαση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Κούν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Κάλλας. Νομίζω ότι πραγματικά είναι συναισθηματικά φορτισμένο το απόψινό θέμα και η ασφάλεια των πτήσεων είναι το πρώτο και θεμελιώδες δικαίωμα των επιβατών. Γι' αυτό ήταν σωστό ότι το Κοινοβούλιο τότε μαζί με την Κομισιόν και το Συμβούλιο ε, συνέστησαν μια ομάδα εργασίας που μπόρεσε να εργαστεί ανεξάρτητα από μέλη των Επιτροπών Ασφαλείας των Κρατών Μελών, από εθνικές αρχές ασφαλείας, με πιλότους και προσωπικό πληρώματα που παρουσίασαν την πείρα τους. Και τώρα υπάρχουν 15 ε, ε, αποτελέσματα ε, σχετικά με το, τους χρόνους πτήσεων. Επίσης από 11 και 45 ώρες ε, μείωσαν το χρόνο στις 11 ώρες στη νυχτερινή πτήση. Επίσης προβλέπουν και διαχείριση της κόπωσης ούτως ώστε να έχουν σωστή η ανάπαυση, οι πιλότοι και κατά τη διάρκεια των πτήσεων των διπυρωτικών, γιατί αυτές είναι μεγάλες πτήσεις που ξεπερνούν το 11ωρο, ε, υπάρχουν ε, διατάξεις για να μπορούν να ξεκουράζονται. Και πολλά ακόμη στοιχεία έχουν συμπεριληφθεί θετικά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά πρέπει να τα λάβουμε όπως τους αξίζει υπόψη. Ε, ορισμένοι επιμένουν ότι η νυχτερινή διάρκεια στα 10 ή 11 ώρες πρέπει να ρυθμιστεί. Ο Επίτροπος Κάλλας μίλησε για 18 ώρες τη βδομάδα. Το, ε, ε, ε, ε, έχουν διαπραγματευτεί και οτιδήποτε υπερβαίνει αυτό το όριο θα ε, καλύπτεται από ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου. Γι' αυτό το ψήφισμα το δικό σας δεν πρέπει να υποστηριχθεί. Θέλουμε τώρα να υπάρχουν διατάξεις για την ασφάλεια των πτήσεων. Θα πρέπει ελάχιστα πρότυπα να εναρμονιστούν ώστε όλοι οι επιβάτες στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό να ταξιδεύουν με τις ίδιες συνθήκες ασφαλείας. Ευχαριστώ. Δέχεστε μπλε κάρτα, κύριε Κούν, από τον κύριο Κράμερ. Ξέρετε συνάδελφε ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μετά από έρευνες απεφάνθη ότι η ΕΑΖΑ είναι η καλύτερη ομάδα λόμπι για τις αεροπορικές μεταφορές στην Ευρώπη πάνω από όλες τις άλλες. Επιβεβαιώνεται αυτό. Επιβεβαιώνεται και ε, επίσης επειδή 30 δις ευρώ παίρνουν από το φορολογούμενο οι αεροπορικές εταιρείε γιατί ε, ε, για τις διεθνείς πτήσεις δεν πληρώνουν φόρο κυροζήνης και ΦΠΑ. αυτά όλα είναι ε, ε, διευκολύνσεις που τους πρόσφερε η Άζα. Τι λέτε εσείς. Καλά, ε, κύριε Κράμερ, ξέρω την πολιτική σας επιχειρηματολογία που τώρα την επεκτείνεται στον φόρο κυροζήνης κλπ. Η ΕΑΖΑ είναι Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας που δεν επηρεάζεται από πολιτικούς ούτε από οικονομικά συμφέροντα. Γιατί αυτό θα μπορούσατε να το πείτε και για άλλες ε, υπηρεσίες ασφαλείας ε, στην Αγγλία ή στη Γερμανία που θα μπορούσατε ε, να πείτε να, να, υπονοήσετε ότι ε, ε, εξυπηρετούν οικονομικά συμφέροντα. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και πραγματικά απορρίπτω αυτή την άποψη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπένιον. Ευχαριστώ. Δεν ε, ήταν ε, ο ευκολότερος από τους φακέλους να κατανοήσουμε αυτός και είναι ένα θέμα με το οποίο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για την απόφαση που θα λάβουμε, γιατί ακούσαμε ότι κοιμούνται οι πιλότοι στην ώρα υπηρεσία τους και <laughs> μάλιστα κανείς δεν θέλει, ειδικά εμείς που είμαστε και συχνοί ε, ταξιδιώτες. Αυτή τη στιγμή το να έχουμε διαφορετικούς κανόνες στα κράτη-μέλη δεν είναι ασφαλές το για τους επιβάτες, το για τους πιλότους, το για τα πληρώματα. Αυτοί οι κανόνες δημιουργούν παραθυράκια όπως ε, για τους ε, χρόνους ξεκούρασης, ανάπαυσης Τώρα, αν δεν κάνουμε κάτι, αυτό σημαίνει ότι θα παραμείνουν αυτά τα παραθυράκια στο Ενωμένο Βασίλειο. Δεν ε, έχουμε κανόνες για ε, τις διαφορετικές ε, ώρες και Επίσης, δεν μπορούμε να αλλάξουμε μόνο δύο ή τρία σημεία χωρίς να δούμε το σύνολο. δεν, θα πρέπει ε, να δούμε ποιες ε, είναι και οι επιστημονικές αποδείξεις και φυσικά εξελίσσονται οι επιστημονικές αποδείξεις ε, και γι' αυτό η αναθεώρηση σε τρία χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντική και για την ασφάλεια των επιβατών αλλά και του πληρώματος και των πιλότων όμως θέλουμε σήμερα αυτούς τους κανόνες για να δυσφαλίσουμε ότι υπάρχει ασφάλεια στην αεροπλοεία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Λιχτενμπέργκερ για δύο λεπτά. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, μας παρουσιάσατε τέσσερα σημεία τα οποία εν μέρει στηρίζονται σε μία ρύθμιση, μελλοντική ρύθμιση, που κατά τις διαβουλεύσεις της, ε, της δεν είχαν υποβληθεί. Να σας εμπιστευθούμε. Ε, μου φαίνεται ότι είναι λίγο υπερβολικό. Στο βαθμό που δεν υπάρχουν διευκρινήσεις και προτάσεις σχετικά με το πώς θα είναι στην πράξη το σύστημα. Δεν μπορείτε να περιμένετε από μας να ε, βασιστούμε μόνο στο λόγο σας ε, όταν παρουσιάσατε εν παρόδο κάποια θέματα που αφορούν βελτιωτικές προτάσεις. Στο βαθμό που δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορούμε να τα συζητούμε. Δεν εκπλήσει το γεγονός ότι ε, υπάρχει τέτοια συναισθηματική φόρτιση στο θέμα αυτό. Ε, τρία θέματα θέλω να προσθέσω. Γιατί για αυτοκίνητα και τα φορτηγά έχουμε πιο αυστηρούς κανόνες ε, από ό,τι για τις ε, αεροπορικές εταιρείες. Γιατί γίνονται δεκτές ε, και παρατίθενται οι μελέτες που ε, τάσσονται υπέρ των αεροπορικών εταιριών και οι άλλες όχι. Και γιατί χαίρονται τόσο πολύ με την πρότασή σας οι αεροπορικές εταιρείες όπως χάρηκαν και για, την για το νομοθέτημα για τα δικαιώματα των ε, επιβατών. Ε, η διάρκεια η εργασίας, ο χρόνος εργασίας, ε, η νυχτερινή εργασία είναι ένα μεγάλο θέμα. Έχει εξεταστεί πολύ και το αποτέλεσμα ε, των μελετών είναι ότι αυξάνονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια αν αγνοείτε τα πορίσματα αυτών των μελετών, κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι ακολουθείτε μια πολύ επικίνδυνη οδό. Εμείς θα πρέπει να ε, τεκμηριώσουμε ότι δρούμε για το συμφέρον των επιβατών, των πολιτών μας και όχι ε, υπέρ κάποιων ε, ομάδων στη βιομηχανία. Δέχεστε από τον κύριο Λάιχτφριντ μπλε κάρτα κυρία Λίχτενμπέργκερ. Ναι, ο κύριε Λάιχτφριντ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Λίχτενμπέργκερ, με αυτή την ευκαιρία θέλω να σας συγχαρώ γιατί Νομίζω ότι το πράσινο ψήφισμα ήταν εκείνο που έδωσε το έναυσμα για να ε, μπουν σε κίνηση κάποιες εξελίξεις που τις θέλαμε και εμείς τότε είχαμε συμφωνήσει. Ε, ήταν σωστό αυτό. Εφόσον τώρα ξεκινάει μια διαδικασία, τι ε, πιστεύετε ότι πρέπει τουλάχιστον να γίνει για να συμφωνήσετε κι εσείς. Ε, αυτό θα πρέπει να το επεξεργαστούμε. Αν τα αποτελέσματα της επιστήμης ε, ληφθούν υπόψη στην ολότητά τους, εν προκειμένου θα συμφωνήσω κι εγώ. Αλλά όταν εξακολουθούμε να αθρίζουμε την εργασία και τη διαθεσιμότητα, το stand-by για να και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη άλλες παραμέτρους δεν μπορώ να συμφωνήσω. Ε, στο βαθμό που προαιρετικά επιτρέπεται κάποια κράτη να ε, έχουν βελτιωμένες προδιαγραφές δεν μπορώ να συμφωνήσω. Στο βαθμό που θα υπάρξουν σαφείς και μονοσήμαντες προτάσεις δεν θα έχω πρόβλημα. Γραπτός όμως, όχι υποσχέσεις εδώ στην Ολομέλεια και όχι γενικολογίες. Αυτά δεν μου αρκούν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Κόχ Τίτερ Λέμπρεχτ. Α, όχι, συγγνώμη, ε, λάθος έκανα, λέει ο πρόεδρος. Ε, η κυρία Ενίν, για ένα λεπτό. Ο κύριος Ενίν. Ευχαριστώ. Ε, η ασφάλεια είναι μεγαλύτερη δύναμη των αέριων μεταφορών. Ε, χάρη σε αυτό, ο αέριο μεταφορέ είναι οι πιο σίγουρε ε, στον κόσμο. Χιλιάδε άνδρε και γυναίκε έχουν πάρα πολύ βαριά καθήκοντα καθημερινά και αν υποχωρήσουμε στον χρόνο καθήκοντο, θα θέσουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού. Σύμφωνα με μία μελέτη το μισό των πιλότων κοιμούνται κατά την ώρα υπηρεσία και όταν ξυπνάνε είδαν ότι και ο δεύτερος πιλότος επίσης κοιμόταν και θα πρέπει να μειώσουμε τους χρόνους για όλου και για τους πιλότους και για τους αεροσυνοδούς και ναι θα πρέπει να περιορίσουμε τους συνδυασμούς χρόνου υπηρεσία και χρόνου αναμονή στο αεροδρόμιο και επίσης ε, όλα αυτά γιατί για να κερδίσουν κάποια χρήματα παραπάνω οι μέτοχοι και τελικά ε, τι θα πρέπει να επιβάλλουμε να μην ε, εργάζονται οι εργαζόμενοι πάνω από 11 ώρες όπως κάναμε και εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόχ, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν Θέλω να ευχαριστήσω τους πιλότες και τα πληρώματα για την υποδειγματική δουλειά τους. Ε, κάνουν το παν για να έχουμε τη μεγαλύτερη ασφάλεια στον κόσμο. Ε, θα πρέπει να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο όμως και γι' αυτό η Επιτροπή ε, εξουσιοδοτήθηκε μαζί με την ΕΑΖΑ να υποβάλουν ένα σχέδιο για τους χρόνους πτήσης, διαθεσιμότητας και ανάπαυσης. Σε τέσσερα χρόνια η ΕΑΣΑ ε, αξιολόγησε πάνω από 40 μελέτες. Δεν είναι τα αποτελέσματα ακριβώς αυτά που ανέμεναν οι πιλότοι, αλλά βελτιώνεται η κατάσταση. Αν απορρίψουμε την πρόταση της Κομισιόν, δεν θα υπάρχει πια πρόταση. Δεν θα έχουν γίνει ούτε μικρά βήματα ε, βελτιωτικά. Θα παραμείνουμε εκεί που βρισκόμαστε. Ε, τώρα όλοι ε, επικρίνουν ορισμένα πρότυπα τα οποία όμως θα συνεχίσουν να υφίστανται. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε τις βελτιώσεις. Δηλαδή να έχουμε για πρώτη φορά ευρωπαϊκά ενιαία πρότυπα τα οποία θα, βρίσκουν, θα βρουν σύμφωνους και, και τα συνδικάτα και τις αεροπορικές εταιρείες. Επίσης, ε, ε, όταν υπάρχουν ε, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις, αυτές δεν επηρεάζονται. Θα υπάρχει το όριο των 13 ώρων την ημέρα που θα μπορεί να μειώνεται ανάλογα με τις συνθήκες της 9. Επίσης η, υπηρεσία στη, τη νύχτα θα είναι από 11.45 στις 11 ώρες. Επίσης Ε, υπάρχει, ε, ε, αυτό σημαίνει μείωση κατά δύο ώρες στην, στο χρόνο υπηρεσίας. Επίσης μετά από 7 ημέρες θα έχει από 36-48 ώρες ανάπαυση και ε, θα είναι βελτιωμένες οι ώρες συνολικά, σε βάση ετήσια δηλαδή. Νομίζω ότι αυτές είναι μεγάλες πρόοδοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοχ. Δέχεστε από τον κύριο Κράμερ μπλε κάρτα. Ορίστε κύριε Κράμερ. Στη ΣΥΠΑ είναι 9 ώρες τη νύχτα και ε, η ΕΠΑ δεν είναι και υπόδειγμα απέναντι στους ε, επιβάτες ε, ούτε πολέμη της βιομηχανίας και παρόλα αυτά έχουν πιο αυστηρά πρότυπα και εσείς θέλετε να μας πείτε ότι τα δικά μας είναι καλύτερα μα πως είναι δυνατόν κύριε Κράμερ ακούστε με οι 11 ώρες ε, είναι για το βράδυ. Εσείς τον μπερδεύετε ίσως και με τις ε, πτήσεις την ημέρα. Η, επίσης ε, η ανάπαυση είναι, πριν από μια πτήση είναι σύστημα καλύτερο και από εκείνο των Αμερικανών. Ο κύριος Λάχτρη τώρα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. είναι λίγο ανοησία αυτό, αυτή η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Είναι λίγο ανόητη. Γιατί από ό,τι φάνηκε δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε όλες τις πλευρές. Μιλήσαμε πριν να ληφθεί αυτή η απόφαση με πολλούς, με τα συνδικάτα, με τη βιομηχανία, με τους πιλότους και στο τέλος ε, υπήρχε κάποια δυσαρέσκεια. Ε, ε, σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν ε, πράγμα που ακούσαμε ε, πολλές φορές κατά τη συζήτηση απόψε. Νομίζω ότι η πρόταση της Κομισιόν πρέπει να τροποποιηθεί και να βελτιωθεί. Πώς? Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Αλλά τώρα η Κομισιόν αρνείται να αλλάξει οτιδήποτε. Γι' αυτό η Επιτροπή Μεταφορών απέρριψε την πρόταση της Κομισιόν. Τώρα ξαφνικά έρχονται οι προτάσεις. Έρχονται όμως ε, μέσα σε μια εβδομάδα, αύριο θα πάρουμε ένα email από την Κομισιόν που θα μας λέει περισσότερες λεπτομέρειες. Μα δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί μέσα σε τρεις-τέσσερις ώρες ε, ε, και μέχρι την αυριανή ψηφοφορία να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι σοβαρή δηλαδή η αντιμετώπιση αυτή. Ενώ η ασφάλεια ε, κατά την πτήση είναι θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Α, μην ψηφίσουμε αύριο. Πρέπει να ε, εξετάσουμε την πρόταση της Κομισιόν και ας αναβάλουμε την ψηφοφορία. Και αν δεν αλλάξει τίποτα ουσιαστικό, τότε πραγματικά πρέπει να πω και εγώ ότι δεν βλέπω κανένα λόγο να την υπερψηφίσω την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντουράν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Bon. Παρακαλώ τι συμβαίνει. Ich weiß nicht, ob ich in politischen Δεν ξέρω αν δεν κατάλαβα κάτι διαδικαστικό, αλλά τα χειροκροτήματα ε, επιτρέπονται και από τα θεωρία. Τι είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα, και οφανές μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Okay, let's continue. Merci, uh, merci. Ας συνεχίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντουρά. Η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να εκφραστούμε σε αυτή την πρόταση δεν δίνει καμία δυνατότητα ούτε διόρθωσης ούτε ενίσχυσης. Και σίγουρα καθόλου με τελευταία στιγμή προτάσεις. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτή η πρόταση αντιπροσωπεύει βελτίωση σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες που ισχύουν αυτή τη στιγμή που είναι ατελείς ε, και ημιτελής. Ε, αυτή η κατάσταση ειναι ατελεις και ημιτελεις αυτη η κατασταση ειναι μη υφιστάμενη συζήτηση. Ε, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Είμαστε πεπισμένοι ότι μετά από 11 ώρες πτήσης, 12,5 ώρες σε περίπτωση αναχώρηση από το απόγευμα, ένας ε, πιλότος είναι σε φάση επαγρύπνησης για να διαχειριστεί οποιασδήποτε λεπτές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι σε μια ε, περίπτωση θα μπορούσε ε, να έχει ε, ε, να μπορούμε να δεχτούμε ότι κάποιες ώρες ανάπναυσης μέσα στο αεροπλάνο θα μπορεί να επιτρέψει ένα πιλότο να, είναι σε κατάσταση που να χειριστεί το, το αεροσκάφος. Θα πρέπει να, κύριε Πρόεδρε, το, κύριε συνάδελφοι, έχουμε, να κάνουμε με την ασφάλεια των πληρώματος και το, ε, επιβατών. Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε λάθος. Αν δεν είμαστε πεπισμένοι για όλες τις καταστάσεις ότι δεν ότι θα είναι πάντα σε ασφάλεια και τα πληρώματα και οι πιλότοι δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να απορρίψουμε αυτή την πρόταση της Κομισιόν και να σας ζητήσουμε κύριε Επίτροπη με, να ξαναστρωθείτε στη δουλειά χωρίς καθυστέρηση και να μας δώσετε συστάσεις, τις τελευταίες συστάσεις από τον επιστημονικό κόσμο. Αυτό, αυτή είναι η δική σας εντολή και το καθήκον σας. Ευχαριστώ. Just now... Και τώρα με συγχωρείτε ήθελα να ζητήσω από όλους που είναι στο βήμα να μην ενοχλούν τους βουλευτές σε αυτή τη συζήτηση γιατί αυτό δεν συνάδει με τους κανόνες μας. Και τώρα θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Ντύρα αν δέχεται μία μπλε κάρτα από την κυρία Άισνερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι Ντουράν, είπα πριν στην ομιλία μου ότι σίγουρα δεν είναι τέλεια η πρόταση. Μπορεί να υπάρξει και καλύτερη βέβαια. Όμως, αν σκεφτούμε ότι αύριο θα εγκριθεί το ψήφισμα και θα απορριφθεί η πρόταση, πιστεύετε ότι αν συμβεί αυτό θα είναι όλα όπως θα θέλετε, τέλεια, και θέλετε πραγματικά από την άλλη πλευρά αύριο αν απορριφθεί η πρόταση να συνεχίσουν να υπάρχουν χειρότερες προδιαγραφές ασφαλείας από αυτές που υπάρχουν στην πρόταση. Ακούστε, για την ασφάλεια δεν έχουμε δικαίωμα στο λάθος και σήμερα η Κομισιόν ε, μας κάνει εδώ μία πρόταση τελευταία στιγμής ε, και μετά αφού αρνηθήκαμε με μία ψηφοφορία και έρχεται εδώ με μία πρόταση, πρέπει να έρθει με μία πρόταση που πρέπει να ικανοποιήσει την ασφάλεια όλων, όχι εμάς τους οικολόγους μόνο. Δηλαδή όταν έρχεστε εδώ και μας λέτε όλα ή τίποτα, όχι δεν δεχόμαστε, ζητάμε από την Κομισιόν να παρουσιάσει σοβαρές προτάσεις σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα για να μπορούμε να κάνουμε μια πραγματική πρόοδο και να υπάρχει εναρμόνιση για όλους και όχι ο καθένας να μπορεί να διατηρήσει την εθνική του κατάσταση γιατί το θέμα των αεροπορικών μεταφορών είναι ένα διασυνοριακό ζήτημα. Ευχαριστώ και τώρα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ο κ. Φερέιρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε. Προσπαθώντας ε, να αποφύγει τη συζήτηση και το δημόσιο έλεγχο, προσποιούμενοι πως ε, δεν ε, είναι ουσιαστικό αυτό που είναι πράγματι ουσιαστικό. Η Κομισιόν θέλει να τροποποιήσει τη νομοθεσία σχετικά με το χρόνο της ισοτοπιλότων και του πληρώματο. Όπως πάντα τυλικούν την πρόταση σε μια ρητορική και λέει ότι θέλει να υπερασπίσει αυτό που θέλει ακριβώς να αμφισβητήσει, δηλαδή την ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών. Η Κομισιόν για μια ακόμη φορά βγάζοντα τη μάσκα δείχνει ποιον υπηρετεί όσο ε, και αν οι εργοδότε ε, του τομέα και μεγάλε μεγάλες εταιρείε θέλουν να μα κάνουν να πιστέψουμε το αντίθετο. Δεν υπερασπίζουν ε, κανείς, δεν υπερασπίζει κανεί την ασφάλεια των ερωματοφορών με επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων όμως η Κομισιόν όπως πάντα αυτούς εξυπηρετεί. δεν αρκεί η συγκέντρωση μονοπωλίων στον τομέα σαν να μην έφτανε η ιδιωτικοποίηση εθνικών μεταφορέων όπως η ΤΑΠΕ στην Πορτοκαλία θέλουν ακόμα περισσότερο να μεγενθύνουν τα κέρδη των κολοσσών των ε, εταιριών αερομεταφορών ε, στις πλάτες των εργαζομένων και της ασφάλειας ε, των επιβατών. Θα δεχτείτε από τον κύριο Ενέν μια μπλε κάρτα, παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Ενέν. Κύριε Φερέιρα, μπορείτε να μου πείτε τι σκέφτεστε για αυτό το κοινοβούλιο που θα αποφασίσει για τη ζωή των ανθρώπων και ε, σε σχέση με το κάποιοι ε, εργαζόμενοι εδώ που έρχονται να παρακολουθήσουν τη συζήτηση, να χειροκροτούν. Κύριε Φερέιρα, όπως ε, είπα... Εδώ έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ποια συμφέρονται περασπίση κομισιών, αλλά όχι μόνο κομισιών, αλλά δυστυχώ και η πλειοψηφία αυτού του κοινοβουλίου. Εδώ σε αυτή την ε, συζήτηση ε, δεν ε, συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, αλλά Σίγουρα αν προχωρήσει αυτή η πρόταση θα έχει και τη δική μας αντίθεση εδώ, αλλά θα υπάρξει και αγώνας των εργαζομένων σε διάφορες χώρες κατά της πρότασης αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙΑΗ. Για ένα λεπτό, κύριο Thank you. I will use the cryptic language which will only... Ευχαριστώ. Θα χρησιμοποιήσω μια κρυπτική γλώσσα την οποία καταλαβαίνει μόνο ο Επίτροπος. Έχουμε πιλότους, έχουμε αεροσκάφη, αερομεταφορείς και παίρνουμε διαφορετικές απαντήσεις ανάλογα με την κάθε άποψη. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει ότι οι εταιρείες κάνουν το σωστό και ότι οι εργαζόμενοι ίσως να κάνουν κάτι λάθος. Για τους οδηγούς δώσαμε βραχύτερους χρόνους απασχόλησης. Ε, η Κομισιόν πιστεύει ότι είναι πιο εύκολο στα αεροπλάνα παρά στα φορτηγά. Ίσως να μην είναι σωστό να ρυθμίζουμε τους πιλότους με τρόπο που να μην αποδέχονται. Γι' αυτό προσβλέπω στην αυριανή ψηφοφορία. Βλέπω ότι το υπάρχει ενδιαφέρον στο θέμα. Θέλω να επιστρέψω στο σπίτι μου με ασφάλεια, με έναν ευχισμένο πιλότο. Δεν θα ε, θα ήθελα με τα χαρά να κάθομαι δίπλα σε έναν ευτυχισμένο επίτροπο. Σας ευχαριστώ. Πάμε να ομιλητή ο κύριος Πάσκα. Κύριε Επίτροπε, πριν από ένα μήνα η μια Βρετανική εφημερίδα μας ενημέρωσε για το ατύχημα ενός ε, Airbus που ε, αντιμετώπισε πρόβλημα διότι ε, χρησιμοποιεί το ο αυτόματος πιλότος επειδή κοιμούνται και οι δύο πιλότοι λόγω υπερκόπωσης. Για ε, λόγους ε, ε, ασφαλείας θα πρέπει να λάβουμε πολύ στα σοβαρά σαν μια κραυγή βοηθεία στο συμβάν αυτό. Ε, πρέπει λοιπόν να ε, λάβουμε υπόψη μας το 10 δεκάωρο και το οκτάωρο άθροισμα 18 ώρων και να το προωθήσουμε. Ε, παραπέμπω άλλωστε και σε επιστημονικά πορίσματα θα πρέπει να βοηθήσουμε και να συνεργαστούμε με τους πιλότους προς το συμφέρον των επιβατών μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να διορθώσω τον τελευταίο μιλητή γιατί η πληροφορία που παρουσίασε εδώ είναι λάθος. Δεν ε, ήταν αυτά τα στοιχεία όταν τα εξέτασε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και νομίζω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, έχουμε από τις ασφαλέστερες ε, αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο. Δεν πρέπει λοιπόν να ε, υπάρχουν παραπληροφορήσεις και παραερμηνίες. Μπορεί να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε στο τι ιδέων γενέσθε. Όμως ε, θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Πιστεύω ότι οι παρεμβάσεις ορισμένων συναδέλφων είναι αντιεπαγγελματικές ε, και ε, Αν δεν είναι αντικειμενικοί, ίσως δεν θα έπρεπε να παίρνουν μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Και τώρα ο Επίτροπος Κάλλας. Α, συγγνώμη, τον κύριο Πάσκα ξέχασα. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι δεν κατάλαβα αυτά που είπατε. Εγώ παρέθεσα επίσημε πληροφορίες από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης και υποθέτω ότι και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας γνωρίζει και συμφωνεί με αυτήν την πληροφορία, δεν τη διέψευσε. Κυρία Σρόιντερ, θέλω να αναφερθώ σε μια επιστολή που έλαβα από εσάς. Εκεί χαρακτηρίζεται την απόφαση της Επιτροπής επί της ουσίας ως παρεξήγηση ε, η οποία στηρίχθηκε σε παραπληροφόρηση από τα ΜΜΕ. Εσείς ε, πώς είναι δυνατόν να ε, ε, παραμορφώνεται έτσι την απόφαση της επίσημης αρμόδιας καθήλυν επιτροπής. Ε, επίσης ε, αναφέρεται και μία επιστολή από τα λόμπι. Ε, εσείς για αυτή τη δραστηριότητα λόμπι τι παίρνετε. Νομίζω ότι όταν ε, συζητάμε το ενδεχόμενο ε, αναθεώρησης μιας απόφασης θα πρέπει να ρωτήσω κι εγώ εάν η απόφαση αυτή στηρίζεται στο, στα δικαιώματα των επιβατών. Ε, τελευταίος ομιλητής ο κύριος Σίμψον. Πρόεδρε, παίρνω το λόγο από τη διαδικασία Κατσιδιάη, γιατί αυτό που με ανησυχεί εδώ είναι ότι υπάρχει κάποια ρεκτηρική από ορισμένου συναδελφού που δείχνει ότι όχι μόνο δεν εμπιστεύονται την ΕΑΣΑ, αλλά και τι δικέ του ρυθμιστικέ αρχέ ασφαλεία. Ε, άκουσα κάποιου να λένε για έλλειψη ασφάλεια, ότι μπαίνουν σε κίνδυνο οι επιβάτε. Το άκουσα αυτό από διάφορε εθνικότητε ε, και το γεγονός παραμένει ότι κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή υποστήριξε αυτή την πρόταση και η γερμανική και η βαλγική και η ισπανική όλες οι ρυθμιστικές αρχές υποστήριξαν αυτό το συγκεκριμένο κανονισμό. Πρέπει λοιπόν να πω ότι υπάρχει κάποια ανησυχία εδώ σε σχέση με την παραπληροφόρηση που κυκλοφορεί και σε σχέση με τους δύο πιλότους. Αυτά που θα έλεγα στο συνάδελφο από τη Σλοβακία, θα έλεγα μην πιστεύεις καταρχήν τίποτα από όλα αυτά που βλέπεις στο βρετανικό τύπο. Καταρχήν και δεύτερον αποφασίστηκε ότι αυτό που είχε υποθεί δεν ήταν σωστό και το είπε ε, η αρχή της ενέργειας κυκλοφορίας. Και σε σχέση με το λόμπινγκ μπορώ να πω ότι ε, αεροπορικές εταιρείε τη Ευρώπη ε, ήρθαν σε μένα να κάνουν λόγο περισσότερο από όλου για πολλά χρόνια. Όμως για το θέμα αυτό πρέπει να πω ότι είχα περισσότερο λόμπι από τα συνδικάτα και κυρίως από τους πιλότους από ό,τι από τις αεροπορικές εταιρείες. Τώρα αυτό μπορείτε να το εξολογήσετε όπως θέλετε, αλλά το λόμπι ήταν ε, έντονο, ήταν ισχυρό και Ας μην ξεκινήσουμε τώρα να μιλάμε για το λόμπι από τις αεροπορικές εταιρείες, γιατί έγινε και από τις δύο πλευρές, ένθεν και ένθεν. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο τελευταίος ομιλητής. Ε, κύριε Κράμερ, έχετε μιλήσει τρεις φορές, δεν είναι δυνατόν να σας ξαναδώσω το λόγο. Και τώρα ο κύριος Επίτροπος για το συμπέρασμα. Κυρίε και κύριοι, Περιμέναμε όλη τη δική σας απόφαση αύριο. Ένα πράγμα να πω μόνο, ότι δεν εκτίμησα ποτέ ε, αυτό που ελέγχθη σχετικά με το λόμπινγκ στον πολιτικό λόγο και μένα μας σε πίεση από τα συνδικάτα και όχι από τους αεροπεταφορείς. Αλλά αν θυμάστε Κατά τη διάρκεια της τελευταίας περίοδου δημιουργήσαμε μια πρωτοβουλία διαφάνειας και ε, κάποιοι εκπρόσωποι ενδιαφερόμενοι ε, καταχωρήθηκαν. Έχουμε 5.700 ε, καταχωρήσεις συμμετεχόντων σε αυτό το Μητρό. Θα πρέπει να δούμε αυτές τις δραστηριότητες lobbying Υπάρχουν αρκετά σχόλια, αλλά σχετικά με αυτό το θέμα τώρα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτός ο πίνακας δεν πρέπει να είναι για πολιτική λήψη απόφασης. Δεν μπορώ εγώ να αποφασίσω τι σημαίνει 4, 45, 10, 45, 10, 15, 10, 30 και αυτό αυτές είναι, αυτή είναι η χρόνια ανάπαυση ανάμεσα στους χρόνους ε, υπηρεσίας. Αυτά πρέπει να παραμείνουν στα χέρια των ειδικών. Και αν απορρίψετε αυτή την πρόταση, εγώ σίγουρα μπορώ να την ε, στείλω πίσω στην ΕΑΣΑ, ο οποίος είναι ένας οργανισμός με μεγάλη φήμη σε θέματα ασφάλειας της αεροπορίας που αναγνωρίστηκε επανειλημμένος. Τώρα, σχετικά με αυτούς τους πιλότους που αποκοιμούνται εν πτήση και ε, ελέγξαμε ότι ήταν λάθος, όπως είπε και η κυρία Φώστερ. Ε, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Ναι, επιτρέπεται να κοιμηθούν. Είναι μέσα στον κανονισμό. Υπάρχει αυτόματος πιλότος σε μεγάλη διάρκεια πτήσης. Είναι περίοδοι κατά τις οποίες ε, μένουν άγρυπνοι και περίοδοι κατά τις οποίες δικαιούνται να κοιμηθούν. Δεν πρέπει να δημιουργούμε την εντύπωση ότι αν κάποιος πιλότος ή ένας πιλότος ε, κοιμάται, τότε σίγουρα ε, το, το αεροπλάνο είναι εντελώς ακυβέρνητο. Υπάρχει μια διαδικασία για τεχνικές τροπολογίες για την αποφυγή λαθών ασφάλειας μετά από κάθε ατύχημα και πρέπει να πω ότι η Ευρώπη είναι η πιο ασφαλής ζώνη πτήσεων. Ε, τουλάχιστον το 2012 δεν έχουμε επιδείνωση των επιπέδων ασφάλειας ε, αεροπορίας. Αυτά λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η πρόταση είναι μια βελτίωση σε σύγκριση με την φυστάμενη κατάσταση. Αλλά όπως είπα, θα περιμένω με ανυπορμονησία την αποφασή σας και απομένουν ε, τα υπόλοιπα στους εμπειρογνώμονες. Τώρα, εκ μέρους της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, θα ήθελα να ζητήσω τα τελευταία λόγια του κυρίου Ελκαντράουι. Eh, eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για αυτή τη συζήτηση. Σίγουρα η ασφάλεια στον τομέα της, ε, των ερωμεταφορών είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλους. Κύριε Κράμερ, είναι αλήθεια ότι εσείς ε, έχετε την τάση να ταυτίζετε όσους πρόκειται να υπερψηφίσουμε αυτό το νομοθέτημα είναι σαν να είμαστε κατά της ασφάλειας. Όμως, ε, αν ε, ψηφίσουμε το δικό σας ε, κείμενο, τότε θα μείνουμε στις 11 ώρες και 45, ενώ η σημερινή πρόταση είναι 11 ώρες. Τη σημερινή πρόταση λέει ότι ο συνολικός χρόνος πτήσεων σε όλο το χρόνο δεν θα είναι πάνω από 1.300 ώρες πτήσης ή πάνω από χίλιες ώρες ε, συνολικά. Όλοι αυτοί οι κανόνες αυξάνουν την ασφάλεια των εργαζομένων ε, ή των πιλότων, αν θέλετε. Και για να κλείσω μπορώ να σας πω ότι πρέπει να αποφύγουμε την εξής παρεξήγηση, αυτή δηλαδή τη σύγκριση που γίνεται μονίμα μεταξύ των εθνικών κανόνων και της συνήθους πρακτικής που πολλές φορές είναι καλύτερη. Υπάρχουν συλλογές συμβάσεις που ισχύουν και θα συνεχίσουν να ισχύουν. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί που, άνθρωποι που δεν έχουν αυτή την κοινωνική προστασία που φοβούνται κάποιοι ότι θα χάσουν και μάλιστα αδίκως φοβούνται και αναφέρομαι στα πληρώματα σε εταιρείε low cost που με αυτή τη σημερινή πρόταση θα έχουν πολύ μεγαλύτερη προστασία από τη σήμερα. Εγώ, ως εισηγητής ε, της Επιτροπολογίας πρέπει να πω ότι εγώ δεν θα υποστηρίξω την πρόταση ψηφίσματος, αλλά όλοι είμαστε ελεύθεροι και φυσικά θα δούμε και τι θα αποφασίσει η Ολομέλεια. Κύριε Κράμερ. Να μου πείτε γιατί ο κύριος Ελκαντράουι μιλάει εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και εκφράζει την προσωπική του γνώμη και όχι την ε, ε, άποψη της Επιτροπής η οποία με αποτέλεσμα 21 προς 13 τάχθηκε υπέρ του ψηφίσματός μας. Ακούστε, ήταν ε, συμφωνία. ο κύριος Μπράιεν Σίμψον συμφώνησε Uh, Έχω μια πρόταση